Let's start, colleagues. Uh, the next point on the agenda is the presentation of the annual report Συνάδελφοι, έχουμε τώρα την ετήσια έκθεση για το 2018 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ο κύριος Μπουταρέλη θα μας μιλήσει, τον οποίον καλωσορίζω. Έχουμε λοιπόν την ετήσια έκθεση της υφιστάμενης εντολής του επόπτη προκειμένου να έχουμε επίσημη και συνολική ενημέρωση για θέματα προστασίας δεδομένων, διαλειτουργικότητα, οδηγία ψηφιακού περιεχομένου, privacy κτλ. Ο επόπτης προετοιμάζει και προς την γραμματεία και την πρώην ομάδα εργασίας ε, εν ώψη της θέσης ενισχύ του GDPR έχει το λόγο ο κύριος Μπουταρέλη για 15 λεπτά σας παρακαλώ. Good morning everybody. Thank you, Madam Chair, for uh, this. Σας ευχαριστούμε, ε, Πρόεδρε, για την παρουσίαση αυτή, για τα καλά σας λόγια. Είναι τιμή για μένα που έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την έκθεσή μας για το 2017. Είναι 14η ετήσια έκθεσή μας ε, ε, και σημαίνει τρόπον την το τέλος μιας εποχής. Διότι όταν θα έρθω για την έκθεση του 2018 δεν θα μιλήσω μόνο για τις δραστηριότητες του επόπτη αλλά και για τη γραμματεία ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας των Δεδομένων όπως σωστά είπατε. Αφιερώσαμε με πολλή ενέργεια για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το νέο οργανό, αυτό το νέο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει από την πρώτη μέρα κιόλας ό,τι χρειάζεται για να προσφέρει άριστες σε παγκόσμιο επίπεδο υπηρεσίες ε, στα μεμονωμένα άτομα ε, και ε, θα βασιστούμε φυσικά στο συναδελφικό πνεύμα και στην καλή βούληση των μελών του Συμβουλίου. Θα δούμε σε διασυνοριακές περιπτώσεις με ποιο τρόπο μπορούμε να παράσουμε συγκεκριμένα συγκεκριμένε συμβουλέ όταν γίνονται οι έλεγχοι. Φυσικά θα επιβληθούν και κυρώσει και θα φανούν οι πολιτισμικέ διαφορέ ανάμεσα στους ε, διαφορου νομοθέτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω ε, θα πρέπει να μιλάμε με ενιαία φωνή, κυρίως ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις για τη χρήση κάποιων προσωπικών δεδομένων ε, για το micro-targeting ε, και την επιγραμμική τους ε, επεξεργασία. Ε, για την, στη ψηφιακή εποχή τώρα ολοκληρώνεται ο κύκλος, αυτός ο ατελείωτος ο κύκλος μεταρρυθμίσεων. Ε, συζητήθηκε με προσοχή αυτό το νομοθέτημα και αποφασίστηκε στο Κοινοβούλιο και θα δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί και τι αποτελέσματα θα έχει ε, σε αυτούς που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή. Ε, ακούγεται σαν κλεισέ, αλλά μπορώ να σας πω ότι η, για τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα είναι ένα ε, ζήτημα που έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, χρειαζόμαστε ε, κατευθυντήριες γραμμές και εμείς, γιατί ξέρετε σε σχέση με ε, μεγαλύτερους οργανισμούς ε, δεν έχουμε έτοιμο προγράμμα για διαχείριση κινδύνων ε, κτλ. Ε, όμως ε, μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί αληθείς οι προβλέψεις μας. πριν από δύο χρόνια μας είδαν με κάποιους ενδιασμούς όταν, είπαμε, όταν προβλέψαμε τις τάσεις των νέων τεχνολογιών. Όμως εμείς τονίσαμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ε, χέγγυα και ασφαλείας που όχι γραφειοκρατία μόνο, το ώστε είναι αποτελεσματική η προστασία των δεδομένων. Επίση, ε, συζητήκαμε ότι ο Γενικό Οργανισμό για την Προστασία των Ατομικών Δεδομένων καλό είναι, αλλά δεν επαρκεί. Και σε μια συγκεντρωμένη αγορά, ε, με του γίγαντε ε, των προσωπικών δεδομένων και το, και το κεκαλυμμένο tracking από τι μηχανέ αναζήτηση, όπω είδαμε από την τελευταία περίπτωση που αποκαλύφθηκε από τον αναλυτή αναλυτή του Κέμπριτζ ε, αποδείχθηκαν ε, αληθείς οι προβλέψεις μας. Ε, και ευχαριστούμε κυρία Γκόμες γιατί ζητήσατε στο στο ενδιαφέρον ψήφισμά σας για τα big data πέρυσι ακριβώς αυτή την ίδια προσέγγιση και μιλάμε για την προστασία την ιδιωτική προσωπικότητα των προσωπικών δεδομένων. να Αγωνιζόμαστε να διαδειχθεί σε προτεραιότητα αυτό το ζήτημα και φυσικά ο θεματοφύλακας είναι το Κοινοβούλιο και έτσι θα έπρεπε να είναι. Θα ήθελα να ε, ζητήσω από τον συνάδελφο Βιουσαρόφσκι να συνεχίσει να δίνει επιστημονικέ συμβουλές στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να δρούμε μετά κατόπιν οδηγιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μετά την θέση εφαρμογή του κανονισμού θα εξασφαλίσουμε τη συνεργεία ανάμεσα στις δικές μας συμβουλές και στη δουλειά που θα κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα είμαστε ενεργό ε, φυσικά του Συμβουλίου. Ε, το Κοινοβούλιο μπορεί να στραφεί σε εμάς για να λαμβάνει ταχαίως επιστημονικές συμβουλές, ε, κυρίως όταν επηρεάζεται η προστασία των δεδομένων, την εφαρμογή και τη χρήση νέων τεχνολογιών. <clears throat> Επειδή μιλάμε για την προστασία των δεδομένων, ήδη από σήμερα θα δείτε στη διεθνή ε, διάσκεψη όλων των επιτρόπων για την προστασία των δεδομένων που θα λάβει η χώρα στις 22 με 25 Οκτωβρίου εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αν θέλετε, για την προστασία ε, των ατομικών ε, δεδομένων. Όχι ότι θα ε, ε, ανταγωνιστούμε ή δε άμυλα. Θα υπάρχει και με κοινό στόχο την προστασία των δεδομένων. Και επειδή είστε ιδιαίτερα προοδευτικός νομοθέτης ε, και βάζετε στην καρδιά του δικαίου τα συμφέροντα του Συνθισμένων συνηθισμένων πολιτών. Θα συνεργαστούμε μαζί σας ε, για το θέμα του κώδικα διοντολογίας, αλλά όχι μόνο με τους συνήθηση υπόπτους. Ε, θα φέρουμε ειδικού ε, για αυτά τα ζητήματα και στο Στρασβούργο θα αναδειχθεί αυτή η πλατφόρμα για την ε, προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων, πέρυσι συνεργαστήκα μαζί σας και με το Συμβουλίο ε, για την πρόταση οδηγίας για το ψηφιακό περιεχόμενο. Ο, ο φόβος ήταν ότι θα υπονομευθεί ο βασικός κανονισμός προστασίας των δεδομένων. Και όπως και για τις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων, Δεν πρέπει να υπάρχουν ε, ε, κενά τα οποία θα θέτουν εν κινδύνο τα τοπικά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες. Ε, ε, δημοσίευσα μια έκθεση για την επιγραμμική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ε, χθε, ε, γιατί, διότι η ουσιακή κοινότητα θεώρησε ότι όλη αυτή η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση για τα fake news, πλαστέ ειδήσει, το λόγο μίσου, το micro-targeting, παραγνωρίζει τη σημασία ενό σημαντικού ζητήματος, παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, δεν υπάρχει έλεγχο, δεν υπάρχει ανάληψη ευθυνών, ε, όταν ε, διάφοροι φορείς παρακολουθούν διαρκώς ε, τις δραστηριότητες τους. Οπότε να υπάρχει συμμόρφωση με την ουσιακή νομοθεσία για να σταματήσει αυτή η επιγραμμική εξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Πριν από 10 χρόνια το ε, κατέρευσε λόγω έλλειψης, ανάληψης ευθυνών ε, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω εκατομμυρίων μικροαποφέσεων και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ρήξης ακριβώς με το ψηφιακό ε, παγκόσμιο σύστημα επηρεάζονται άμεσα οι δημοκρατίες μας ε, κυρίως τώρα που πλησιάζουν και οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Κάτι τελευταίο για τις ε, πρώτες δραστηριότητες μας ε, και για το, ε, τη μορφή που παίρνει ο κανονισμός 45-2001. Όπως και εσείς, ε, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δίνει το παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νομοθεσία που εγκρίνει και στον τρόπο που εφαρμόζει αυτά τα νομοθέτηματα. Η ευθυγράμμιση του GDPR θα πρέπει στο μέτρο να ε, προς ε, τα, ε, τις νομικές πράξεις ε, του πρώην τρίτου πυλώνα για την ε, συνεργασία στα, στο τομέα του ποινικού δικαίου. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την ιδέα ένας νόμος για όλα, κυρίως για τα προσωπικά δεδομένα διοικητικού χαρακτήρα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το στόχο της προστασίας των ευρωπαϊκών δεδομένων διατηρώντας τα ιστάμενα πρότυπα αλλά εξασφαλίζοντας και συνοχή και προ προβλεψιμότητα κυρίως για τα υποκείμενα θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο η ε, Europol μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και βεβαίως θα πρέπει ε, οι διάφορες υπηρεσίες ε, να δημιουργήσουν ένα σύστημα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των στοιχείων που έχουν έτσι ώστε όλα να μπουν στην ίδια βάση δεδομένων. Επομένως, διαρκώς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή καθώς επίσης και με θέματα τα οποία σχετίζονται με την ανάλυση των προϊόντων και βεβαίως βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Κοινοβούλιο, το οποίο έχει φέρει ένα σημαντικό ε, βαθμό της ε, ευθύνης για την προστασία των ε, προσωπικών δικαιωμάτων. Έχει γράψει ιστορία ε, το σώμα αυτό και οπωσδήποτε αποτελεί έμπνευση και για τους άλλους ε, σε σχέση δηλαδή με την ευρωπαϊκή προσέγγιση του θέματος. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. μένει ένας χρόνος ε, μέχρι τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές ε, και πραγματικά θα ήθελα να ξέρετε ότι βρισκόμαστε απολύτως στην ε, διάθεσή σας με όλες μας τις δυνάμεις για να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε το έργο που ξεκινήσατε. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν όσον αφορά ε, και το, τον 45-2001 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ε, υπάρχουν πολλές ηλεκτρονικές ε, ανακοινώσεις και βεβαίως ο στόχος είναι να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση, Ένα στόχος ο οποίος δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί. Υπάρχουν ε, μέλη τα οποία βοήθησαν πάρα πολλέ διαδικασίε και τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν θα ξανά είναι υποψήφια στις επόμενε εκλογέ. Η ομάδα Μπένενστη την προηγούμενη εβδομάδα ε, αναγνώρισε ότι υπάρχουν δύο στάδια για την ε, ψηφιακή ζωή. Ε, πρώτον, ότι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθεί η ψηφιακή ευημερία είναι η κεφαλαιοποίηση των στοιχείων. Δεύτερον, ότι μονάχα οι μεγάλες πλατφόρμες μπορούν να βρουν λύσεις. Αυτό δεν είναι σωστό για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και γενικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν είναι δίκαιο για την Ευρώπη, δεν είναι όμως δίκαιο και ε, ε, για τους διάφορους ε, γίγαντες του τομέα αυτή είναι η δικιά σας ε, ε, δουλειά και εσείς θα πρέπει να προστατεύσετε τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή με την οποία με ακούσατε και βεβαίως είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε διευκρινήσεις ή ερωτήσεις. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουταρέλη για αυτήν την τόσο πλήρη τοποθέτησή σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στους ε, ε, βουλευτές. Ε, πρώτα απ' όλα η κυρία Κιάνγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον δόκτωρα Μπουταρέλη για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη διότι το θέμα των ε, ημερών, το οποίο και εσείς άλλωστε αναφερθήκατε, είναι ακριβώς η δεοντολογία στην προστασία των δεδομένων ε, και βλέπουμε ότι έχει εντελώς τσαλακωθεί αυτή ε, η ιδέα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα όσα συνέβησαν με την Cambridge Analytica γιατί εδώ μιλάμε για κατάφορη παραβίαση των δεδομένων ε, και ε, ε, ξεγυμνώνεται η αδιαφάνεια όσον αφορά τη διαφάνεια όσον αφορά συγγνώμη, τα δεδομένα των χρηστών καθώς επίσης και όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Επίσης σχετίζεται εδώ και θέμα των εκλογών και των εκλογικών διαδικασιών άρα δημιουργούνται και προβλήματα όσον αφορά τις δημοργατικές διαδικασίες εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο hate speech, στον λόγο μίσους. Ε, τι μπορεί να γίνει όσον αφορά το θέμα αυτό και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καταστάσεις παρόμοιες με την Cambridge Analytica. Σας ευχαριστώ. κύριος Δίας Νεμέρα έχει Ευχαριστώ τον κύριο Μουταρέλη για την παρουσίαση της εκθέσεώς του. Εχθές σας είδαμε εξ αποστάσεως από την Σοφία. Σόφια. Παρότι εσείς δεν μπορούσατε να μας δείτε βεβαίως. Ήθελα να εκφράσω μία κάποια απορία για το δεύτερο τμήμα της θετικής αποτίμησής σας για την προστασία των δεδομένων στα πλαίσια της Ευρωπόλ. Είπατε ότι α βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά β και σε αυτό αναφέρομαι σχετικά με κάποια διευκρίνηση ή αποσαφήνιση, μιλήσατε για περίοδο τήρησης των δεδομένων και σχετικά θέματα με την ανάλυση. Εγώ θα ήθελα λοιπόν μια περαιτέρω ανάπτυξη επί της ανάλυσης αυτής των δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αγκουστίν. Ο κύριος Λόπες Αγιλάρ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Μπουταρέλη, για τη δουλειά που έχετε κάνει στον επόπτη. Έχουμε μία αλληλουχία σκανδάλων αυτή τη στιγμή που πλήττουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στο δίκαιο. Διότι είναι προφανές ότι τα μονοπόλια που ασκούν οι γιγαντιές επιχειρήσεις του διαδικτύου αποσαθρώνουν τις εγγυήσεις που είχαμε απόλυτα σε θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ο κανονισμός προστασίας δεδομένων που εισάγει μια ενίσχυση σχετικά με τη διόρθωση ή διαγραφή αυτό που αναφέρουμε ως δικαίωμα στη λύθη προκειμένου να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη εκείνα δικαιώματα που αυτή τη στιγμή απειλούνται όσο ποτέ από μεγάλες επιχειρήσεις, από μεγάλα μονοπόλια όπως έλεγα, τα οποία εκφεύγουν του θεσμικού ελέγχου των κρατικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και τελικός επιβολής του δικαίου. Ο γεωλογικός εντοπισμός, ο γεωγραφικός εντοπισμός, η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στην ιδιωτικότητα και την προσωπική ζωή του καθενός που ενέχει το big data θα καταστήσει απολύτως αδρανεί αυτήν την ενίσχυση που εισάγεται μέσω της τροπολογίας στον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Άννα Ευχαριστώ τον κύριο Μπουταρέλη για την παρουσία του. εκτιμώ ακόμα περισσότερο την παρουσία του μια και γνωρίζουμε ότι δεν είναι απόλυτα καλά στην υγεία του. Παρ' όλα αυτά ήρθε. Η υπηρεσία που παρέχεται είναι θεμελιώδους σημασίας και ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον θεωρείτε ότι το GDPR είναι έτοιμο να υλοποιηθεί από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Είχαμε εκπροσώπους εδώ πρόσφατα στο Κοινοβούλιο που μας είπε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι έτοιμες, αλλά οι μικρές και μεσίες πώς το βλέπετε, τι περιμένετε. Βεβαίω και συμμερίζομαι τις ανησυχίες ε, που ανέφερε η Cecil King για την Cambridge Analytical. Ποια θα ήταν η σύστασή σας προς εμάς και τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Γιατί τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα πεδίο κρίσιμης σημασίας. Βλέπουμε και πολύ σημαντικές εξελίξεις στα κρυπτονομίσματα, π.χ. και πώς αυτό υποβοηθεί το ξέπλυμα του χρήματος ή τρομοκρατικές δραστηριότητες. Ακούμε για προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης drones που χρησιμοποιούνται για στρατιωτική και αστική χρήση. Ακούμε για το πρώτο ατύχημα που έγινε κατά πεζού από όχημα χωρίς οδηγό. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι πώς μπορεί να διακυβερνήσει το σύνολο του πλαισίου αυτού και η τελευταία μου ερώτηση είναι η διάδραση του πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων και με το δικό σας οργανισμό επόπτη. Εμείς στην Πορτογαλία έχουμε μια εθνική επιτροπή που συνήθως υποβάλλει πάρα πολύ αξιόλογες γνωμοδοτήσεις προς την κυβέρνηση, καμιά φορά τις υλοποιούν κιόλας. Η εθνική μας αυτή επιτροπή όμως από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να καλύψει αυτό το τεράστιο σκάνδαλο με τις χρυσές βίζα που ενέχονται και πρώην υπουργοί της κυβερνήσεως ε, ο υπουργός εκείνος που αυτή τη στιγμή κατηγορείται είναι υπόδικος, έχει χρησιμοποιήσει μια γνωμοδότηση της Εθνικής μας Επιτροπής Προστασίας Δομένων, επικαλούμενος ακριβώς την προστασία των δομένων, ώστε να μην παραδοθεί ο κατάλογος των πληροφοριών που υπήρχαν στη δικαιοσύνη. Δεν είναι παράλογο αντί να εκπληρώνει το καθήκον της μια εθνική προστασία προστασίας δομένων να χρησιμοποιείται προκειμένου να προστατεύσει ένα σύστημα που είναι διεφθαρμένο. Αυτό θα σας το υποβάλω και γρατώζω με όλα τα έγγραφα που έχω στη διάθεσή μου. Μάλιστα, να ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Μπουταρέλη για την του. Ευχαριστούμε για τη δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρατε ήδη, Πρόεδρε, ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ξεκινήσαμε με την προστασία των δεδομένων, μιλούσαμε για κάποιες εκτυπώσεις, ε, κάποια έντυπα, κάποια τηλεφωνήματα, ίσως και κάποια email. Αλλά η τεχνολογία τρέχει Μιλούμε για το ίντερνετ των πραγμάτων, τα συνδεδε, τις συνδεδεμένες συσκευές κτλ. Και από όλο αυτό το ψηφιακό πλαίσιο αντλούνται δεδομένα από τις συσκευές μας, τις 20 συσκευές, το ψυγείο, το πλυντήριο. Δεδομένα συλλέγονται από παντού. Είναι λοιπόν σημαντικότατο να έχουμε ισχυρούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, αλλά παράλληλα, όπως είπατε και εσείς, χρειαζόμαστε και πρόσθετες ρυθμιστικές πράξεις ή πλαίσια. Και μαζί με την τεχνολογία που τρέχει και καλπάζει προς τα εμπρός, διατρέχουμε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι στο τέλος ένα, ένας μικρός μόνο αριθμός επιχειρήσεων που θα ελέγχει, όλων αυτών των όγκο δεδομένων που θα συλλέγονται. Επηρεάζοντας πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά όχι μόνο. Πολλοί λένε ότι με όλα αυτά τα δεδομένα που μόνο κάποιοι λίγοι φορείς τα χειρίζονται, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία θα απειλείται το ίδιο το σκεπτικό, η ίδια η έννοια της προσωπικής ζωής, γιατί θα έχουμε μπει πλέον στο πεδίο του smart living. Επομένως, πρώτη ερώτηση. Το GDPR θα τεθεί ισχύ το Μάιο, αυτό είναι κοντά. Αλλά η εντύπωσή μου, και ίσως μπορείτε να μας πείτε κάτι, δεν είναι όλοι έτοιμοι να δουλέψουν τους νέους κανόνες. Επίσης, Ποια είναι η άποψή σας για το κατά πόσο στα κράτη-μέλη υπάρχουν επαρκώς καταρτισμένοι ειδικοί, αξιωματικοί, κρατικοί λειτουργοί για να αναλάβουν την προστασία αυτήν. Επί του e-privacy δεν έχουμε επίσημη τοποθέτηση από το Συμβούλιο, αλλά ακούμε ότι κάποια κάποια κράτη-μέλη, κάποιοι φορείς θα ήθελαν ακόμα περισσότερο να αποδυναμώσουν από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μην μιλήσω καν για την τοποθέτηση αυτού εδώ του Κοινοβουλίου. Δουλεύουμε κάπως ε, στα θέματα τα φορολογικά και του ανταγωνισμού, αλλά δεν ξέρω αν έχετε και άλλα εσείς κατά νου, ούτε ξέρω αν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, αλλά έχω την εντύπωση ότι μια και ακούμε και φήμης ότι μεγάλες Επιχειρήσει του διαδικτύου καταβάλουν ε, ε, φορολογική επιβάρυνση 2-3% για τους πολίτες που εκπροσωπώ θα σας πω αυτό είναι γελίο. Δεν καταλαβαίνω καν γιατί έχουμε φορολογίες εξαιρέσεις για αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις του ίντερνετ. Αλλά τέλος πάντων. Μερικές εβδομάδες, πριν από μερικές εβδομάδες μιλούσαμε και για την ε, ασπίδα της ιδιωτικότητα το Privacy Shield, αλλά δεν ξέρω αν έχετε περισσότερα να μας πείτε για το πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Και βεβαίως η κυρία Ένστ Ευχαριστώ πρόεδρε. Πάντοτε χαίρομαι που σας υποδέχομαι όταν σας βλέπω κύριε Μπουταρέλη, εσείς εκπροσωπείτε μια προοδευτική τοποθέτηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία των δεδομένων εμπίπτει σε αυτήν την πολιτική τοποθέτηση. Πριν από λίγους μήνες ήμουν στη Βουλγαρία Έβαλα τα γυαλιά και κοίταζα και λέω ναι, ναι, ναι, σωστά. Όταν μιλάμε για την εφαρμογή του GDPR, και πολλοί υπέδειξαν ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και στη Γερμανία λένε όλοι αμάν αμάν πώς θα εφαρμόσουμε το βασικό κανονισμό ε, και δεν ξέρουμε αν είναι εφικτό όταν μιλάμε κυρίως για μικρές επιχειρήσεις. Ε, γι' αυτό μπορείτε να μας πείτε, έχετε σφαιρική άποψη, η κατάσταση πώς είναι στα κράτη-μέλη, σε ποια κατάσταση ε, βρίσκονται, θα μας βοηθούσατε. αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, σωστά είπατε, πως το ευρωπαϊκό επίπεδο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να καταβάλει προσπάθειες ε, για να παρασχεθεί υψηλή προστασία και δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, για, ε, μόνο για τους δημόσιους φορείς ε, στα κράτη-μέλη και να παραγνωρίζουμε λίγο, να κλείνουμε τα μάτια έστω και λίγο για την κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσείς το ίδιο μας υπενθυμίσατε ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιο καθεστώς ισχύει που να μας εξασφαλίζει προστασία υψηλής ποιότητας. Χάνω και τα λόγια μου, δεν μπορώ να τα πω. Και ξέρετε ότι όταν μιλάμε για τον κανονισμό, ε, ε, ε, ε μήνες ολόκληρους αγωνιζόμαστε ναι, και ήταν σαν το Άγιο Δισκοπότερο αυτός ο κανονισμός. Λοιπόν, ε, όπως και σε άλλου άλλους τομείς, ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί παντού αυτός ο κανονισμός και στους εξωτερικούς οργανισμούς και στου στους ιδιωτικούς φορείς παντού. Κατά τη γνώμη σας, ε, τι πρέπει να κάνουμε για να δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία σε περιπτώσεις ε, που παρεμποδίζεται. Αν και κάτι άλλο, ε, επειδή το αναφέρατε πολλές φορές, μιλήσατε για την διαφορά λέξη generalis και λέξη specialis. Ωραία. Όταν Βασιζόμαστε σε αυτό, ωραία, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο συσχετισμός των δύο. Λοιπόν, ε, αυτός ο συσχετισμός ε, του γενικού, της γενικής και της ειδικής νομοθεσίας, ακριβώς ποιος πρέπει να είναι για να μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα βοηθούσε ε, στη συζήτηση να μας δώσετε κάποιες ιδέες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μπουταρέλη έχει ε, τώρα το λόγο για να απαντήσει. Thank Ευχαριστώ. Με την κυρία Γκέγγε θα αρχίσω. Φέτος, μετά τη σκληρή δουλειά που κάναμε, καταφέραμε εδώ μπροστά. Κάνουμε τη... Θα κάνουμε τη διεθνή συζήτηση για τον κώδικα διοντολογής για τις ε, τε, προηγμένες τεχνολογίες. Η... Ε, Κανόνε ιδιωτικού δικαίου για την προστασία των ε, ατομικών δεδομένων θα έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά αυτό δεν επαρκεί αυτό, διότι λείπουν άλλα δύο κομμάτια του παζλ το e-privacy και η νομοθεσία για τα όργανα και τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αρχίσαμε με την άσκηση του για, για, τα καταπιστεύματα και για τις ε, συγχωνεύσεις και την προστασία των επικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό αναφέρω αναφέρθηκα σε αυτό που δημοσίευσαμε χθε στις ε, πλαστέ ειδήσει, ε, δηλαδή την περίπτωση Cambridge Analytics. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση, διότι με την ε, τεχνητή νοημοσύνη και με τον, ε, τις προηγουμένες τεχνολογίες ε, που εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση ε, της, της, της εξουσίας στα χέρια κάποιων μόνο λιγοστών τεχνολογικών γιγάντων καθιστά απαραίτητη τη νέα νομοθεσία για τα οπτικοακουστικά μέσα και γενικότερα για το τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ε, πως ό,τι είναι τεχνολογικά εφικτό είναι και ευκταίο από πλευράς ήθους. Όχι. Ε, πρέπει να συζητούμε με την κοινότητα των σχεδιαστών, των παραγωγών, των κατασκευαστών, των διανομέων που δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, όμως φέρουν παρόλα αυτά μεγάλο μέρος της ευθύνης. Θεωρούμε ότι η αξιοπρέπεια είναι μια αρχή που δεν γίνεται σεβαστή παρότι προβλέπεται στο πρώτο άρθρο τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στη διεθνή διάσκεψη Ακριβώ μετά την ε, ε, σύσκεψη για την ε, τεχνητή νοημοσύνη θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τι σημαίνει, ποια είναι αυτή η ηθική διάσταση στο πλαίσιο της μεταβιομηχανικής επανάστασης. Ποιο μπορεί να μιλά καν για αρχές διοντολογίας και μπορούμε να μιλάμε για εφαρμοστέα κριτήρια σε παγκόσμιο παγκόσμιο επίπεδο, διότι δεν έχουμε θεσπίσει διεθνή πρότυπα για την προστασία των ατομικών δομέων μέχρι στιγμής. και πώς μπορεί να γίνει αυτό στον τομέα των ηθικών πρωτήτων και δεν δε θέλουμε τώρα φιλοσόφους, επιδημιολόγους, ε, ερευνητές, τους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή για να καταλάβουμε πώς ε, εφαρμόζονται αυτές οι αρχές διατολογίες στι διαφόρους ε, τομείς για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα σε σχέση με το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε αυτή την ολιστική προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων. Πιστεύουμε πως είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η συζήτηση. Δημοσιεύσαμε ήδη την ενδιάμεση έκθεση ε, για τη δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί τον ε, Ιούνιο για τον ε, επόπτη αυτό, για τον Ευρωπαϊκό επόπτη ε, και τον Οκτώβριο αναμένεται η σημαντική συζήτηση αφού ομαδοποιήσουμε όλα τα δεδομένα και δεν θα εμπλάκει μόνο το Κοινοβούλιο αλλά όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διεθνή συζήτηση για τη διοντολογία. Κύριε Δίας μέρα ε, ε, καλά τα είπατε, ναι, ε, με τη Europol αρχίσαμε δύσκολα, ε, είχαμε μεταβατικές κατευθυντήριες γραμμές, προσωρινά εγκρίθηκαν χωρίς να διαβουλευτούν μαζί μας όμως. Μήνες μετά και σε μια σύσκεψη που είχα, με το Διοικητικό Συμβούλιο με καθίχασαν διότι οι πλέον σημαντικέ συστάσει μας όντω είχαν ληφθεί υπόψη. Για την διατήρηση των δεδομένων ξέρουμε πως πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, βασιζόμαστε στην αναγκαιότητα και στην αλογικότητα, κατά περίπτωση να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ανακατηγορία. What? Τι ε, να κάνουμε, πώς μπορούμε να επιτύχουμε την ε, σωστή ισορροπία. Και ταυτόχρονα με την αποστολή της προστασίας των δεδομένων να εντοπίσουμε και τις ε, πλέον πρόσφαρες λύσεις. Αλλά παραμένω αισιόδοξο όχι μόνο ε, γενικότερα για τη στρατηγική, αλλά και για τα επιμέρους ε, σημεία για την ε, διατήρηση των δεδομένων. Ο κανονισμός GDPR για τους γίγαντες της τεχνολογίας. Κύριε Λόπες Αγγιλάρ. Ε, πρώτη φορά υπάρχει μια ξεκάθαρη Δεν μας νοιάζουν οι σερβες, το establishment, τα ε, ε κεντρικά γραφεία των επιχειρήσεων. Εμείς βλέπουμε πού, πού προσφέρονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για την εδαφικότητα. Ε, πρώτη φορά ε, θα έχουμε μία προσέγγιση άσπρο-μαύρο. Δηλαδή, ε, το κανονισμό GDPR θα εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους γίγαντες. ας επιστρέψω το 95 και στο 98. Ε, αυτό το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας 9546 αμφισβητήθηκε λόγω πανικού από αυτούς τους, μεγάλε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που προσπαθούσαν να αναβάλουν ε, την προθεσμία για τον Οκτώβριο του 1998 και τώρα βλέπω η Microsoft, η Google και άλλοι κοινοποιούν την πρόθεσή τους να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του κανονισμού. Καταλαβαίνουν ότι ε, ε, το να κατακαιρματίσουν αυτή την πολιτική ε, ιδιωτικότητα θα ήταν μόνο παρελκυστική συμπεριφορά και πιστεύουν ότι με επιτυχία μπορούν σε παγκόσμιο επίπεδο να εφαρμόσουν αυτά τα πρότυπα. Το θέμα είναι η ικανότητα στην πράξη να είναι αποτελεσματική η δράση. Επίσης, η ικανότητά μας να εκφραζούμε μια ενιαία άποψη και γι' αυτό ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας των Δεδομένων θα έχουμε αυτές τις νέες προσεγγίσεις, αυτές τις νέες αρχές. Συναδελφικό πνεύμα, εξυγχρονισμός, διαφάνεια, λογοδοσία, επιλεκτικότητα ε, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε συνένεση και όχι ε, να στρέφονται πάντοτε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός συνοχής και αν ε, ε, παρακάμψουμε την ε, και μάλλον παγιδευτούμε στην γραφειοκρατία, θα εγκλωβιστούμε για εβδομάδες ολόκληρε. Εμείς θέλουμε να προλάβουμε αυτή την κατάσταση και να μιλάμε, να δρούμε συνενετικά στο μέτρο του δυνατού. Με του tech giants, τώρα τους τεχνολογίες, Νομίζω ότι καταδείξαμε την κοινή μα προσέγγιση. Συγχρονίστε τι προσπάθειε που κάνουμε για την περίπτωση Facebook ε, για την ε, πολιτική ιδιωτικότητα των δεδομένων ε, επίσης στη περίπτωση Microsoft για το cloud, έτσι, για το σύννεφο δεδομένων Microsoft εναντίον FBI και Υπουργείου Εξωτερικών, τον είπα, φάνηκε αυτό και η 25η Μαΐου σίγουρα θα είναι ορόσημο. Πρέπει επίσης ε, ε, στις, ε, με βάση τη αρχή αναλογικότητα να εφαρμοστεί αυτό και μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσει. σήμερα το πρωί και το απόγευμα θα τα πούμε με του συναδέλφου πώ ακριβώ θα εφαρμόσουμε το άρθρο 30. 5. Για εφαρμοστική πρακτική, δηλαδή για το GDPR, αποκλιμακωμένο. Ε, ως προς εξαιρέσεις ε, ε, εξαιρούνται οι επιχειρήσει αυτόματα ή κατά περίπτωση ανάλογα τι κάνουν ως προς την το πόσο ευαίσθητα είναι τα δεδομένα δηλαδή. θα δημοσιεύσουμε γιατί η, η σε ολοκληρώνει σύντομα τις εργασίες της για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα Cambridge Analytics. Ε, δεν είναι καινούργια αυτό το πράγμα, δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια παραβίαση και πριν από μήνες αρχίσαμε σε παγκόσμιο επίπεδο να κάνουμε μια επιστημονική προσεκτική ανάλυση των ε, ρηξικέλευθων τεχνολογιών. Δηλαδή, με ποιο ε, καινοτόμο τρόπο συλλέγονται τα δεδομένα, διατηρούνται, γίνονται παρεκβολές και βγαίνουν από τα συμφραζόμενα τα δεδομένα. Λοιπόν, ε, με τα infonomics και τις διάφορους διάβλους που χρησιμοποιούν για την εξαγωγή πληροφοριών, βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται, πώς χειραγωγούν τα δεδομένα και πώς θα επεξεργάζονται με σκοτεινό τρόπο, εκτός ε, πλαισίου, εκτός ε, συμφραζομένων, ε, χρησιμοποιώντας όχι μόνο λογισμικά για την επεξεργασία των δεδομένων, αλλά δημιουργώντας σε μια ψευδεπίγραφη πραγματικότητα, ούτω ώστε να έχουν το πλεονέκτημα να έρχονται πρώτοι σε επαφή με τους ενδιαφερομένους. Βλέπουμε όπως ένας γιγάντας μπορεί να εφαρμοστεί από 52.000 διαφορετικούς τρόπους για να κάνει profiling του χρήστη, κάτι που είναι αόρατο ε, στο ε, μα το απλού θεατή. Και ε, το μικρόφωνο του υπολογιστή σας, το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε, όλα αυτά δίνουν πληροφορίες και άλλα παραδοσιακά μεν ενδιαφέροντα δε λογισμικά που με αδιαφανή τρόπο οδηγούν σε συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, ε, ε, ε, θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε τη νέα τεχνολογία, να δούμε οι αλγόριθμοι με ποιο τρόπο επιτρέπουν την εντελώς διαφορετική χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν μιλάμε μόνο για την προστασία της προσωπικότητας, για όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνδέονται με την ίδια τη δημοκρατία. Ε, οι προηγούσες έρευνε, όχι μόνο στη ΣΥΠΑ αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις micro-targeting και ε, επιγραμμικής χειραγώγησης ε, δεδομένων, οι χρήστες ε, δίνουν πολύ περισσότερα Και αυτό το, το, το φαινόμενο, συγγνώμη, εντείνεται όταν ε, θεωρούνται πλαστές, ε, πλαστά τα δεδομένα παρά αληθή. Δεν έχουμε... Ε, ε δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε ε, μαγικές προβλέψεις ε, θέλουμε, όμως δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προδικάσουμε το μέλλον, όμως θέλουμε να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, θέλουμε ε, συνενετικά να εκφράζουμε την άποψή μας ε, και να επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε στρατηγική διάσταση του ζητήματος, οπότε γι' αυτό κατά προτεραιότητα αποτινόμαστε σε εσά και σε άλλους που εκπονούν πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να θέσετε και στις συνθήκες εργασίας για τις έρευνες που κάνετε από πλευρά Θα συγχρονίσουμε τις, ε, τις ε, πρωτοβουλίες σας με άλλους ε, συναδέλφους. Σε ποιο σημείο είμαστε για το GPR. Κάποιοι έχουν καθυστερήσει Ε, υπάρχουν θέματα με την ε, γερμανική και αυστριακή νομοθεσία και το τελευταίο σχέδιο, νομοσχέδιο που ενέκρινε ο Ολλανδός ε, νομοθέτης. Ακόμη και στη χώρα μου, σε κάποιες περιοχές, έχουν χάσει την μπάλα λόγω γενικών εκλογών. Και... Υπάρχει ένα σχέδιο, είχα την τιμή να το δω αυτό το προσχέδιο. Δεν μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε, με ικανοποίησε 100% αλλά προσπαθούμε να τους πείσουμε και με παιδαγωγικό τρόπο για ε, χρονικά και για το περιεχόμενο να τους ε, πείσουμε. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε την ε, παρέμβαση των διεθνών νομοθετών για τις απαιτούμενες προσαρμογές να μην παραβιάζουν δηλαδή την ναι, ενωσιακή νομοθεσία, αλλά να ασχολούμαστε με κάποιε αποχρώσεις αμφιλεγόμενε ε, τη ε, κείμενη ε, ενωσιακή νομοθεσία και να ευθύσουμε την προσοχή πρώτα απ' όλα τη ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτές τις περιπτώσει. Εμείς έτοιμοι είμαστε από πλευρά νομοτεχνική, αν θέλετε, αλλά μπορούμε να υποφεληθούμε από την γενική ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου. δημοσιεύσαμε και τη μελέτη οι ε, DPS του επόπτη ε, ε, καταθέσουμε και στα πλαίσια του σχεδίου προπολογισμού για το 2019 στα συναρμόδια όργανα γιατί στην Ευρώπη έχουμε νέες, νέους πορούς αύξηση 24% 2000 Ε, ε, ε, ε, δεν είναι πάρα πολλά σε σχέση με αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά ψίχουλα δηλαδή, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα ε, μέρα, θα με, λιγότερους πόρους. θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιλεκτικοί, να δρομολογήσουμε, να ευθυγραμμίσουμε τις διαδικασίες μας και όπου χρειαστεί να περιμένουμε περισσότερο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 ίσως μέσα σε έξι μήνες και αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα γνωστά φόρα, όπως ας πούμε η ετήσια κοινή συνεδρίαση των ε, Εθνικών και, Ευρωπαϊκών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, ίσως καταφέρουμε, λέω, να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη μία ε, συζήτηση για τον ρόλο που μπορούν να παίξουν και σε εθνικό επίπεδο εντός των πλαισίων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Ε, υπάρχει μία τάση επανακερματισμού, υπάρχει μία τάση έτσι, διαχωρισμού ε, χρησιμοποιώντας ε, και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιώντας κυρίως τις, τροπολου... τις προσθήκες, τροποποιήσεις κλπ. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή ε, προσέγγιση δεν είναι δυνατόν ε, το 2020 να έχουμε ακόμα επόπτες ε, που θα πρέπει να ασχολούνται με αυτές τις νομοθεσίες οι οποίες δεν έχουν σωστά υλοποιηθεί και ενσωματωθεί στο νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών. και για αυτούς που καλή την πίστη θέλουν να εφαρμόσουν τον ε, γενικό κανονισμό αλλά είναι παγιδευμένοι κατά κάποιο τρόπο από τους προηγούμενους ε, κανονισμούς και κανόνες η κατάσταση θα είναι καταστροφική. Επομένως άσχετα από το ε, είδος των συμβιβαστικών λύσεων και συμβιβασμών εγώ αυτό που σας ενθαρρύνω να κάνετε είναι να επιμείνετε έτσι ώστε ο γενικός ε, κανονισμός να ε, υλοποιηθεί ε, σωστά. Επίσης, συμφωνώ με την κυρία Έρστ σχετικά με τον, 45, τον κανονισμό 45-2001 δεν υπάρχει πλέον χώρος για κατακαιρματισμό ας πούμε των διοικητικών ε, δεδομένων. Οι αρχές θα πρέπει να είναι ίδιες. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη ε, κάποια επιχειρησιακά δεδομένα ή για, κάποια, ε, για κάποιες άλλες περιπτώσεις να ε, προβλεφθούν όχι απαραίτητα εξαιρέσεις αλλά οι, ε, προσήκουσες διηγητικές ρυθμίσεις λαμβάνοντας υπόψη μονάχα την ιδιαιτερότητα κάποιων δραστηριοτήτων και στοιχείων. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά. Υπάρχει το κεφάλαιο 8 το οποίο ταυτοποιεί τα στοιχεία αυτά. Και βεβαίως αυτό που βλέπουμε εμείς σαν ενδεχόμενη λύση και αναφερθήκατε στο συσχετισμό ανάμεσα στο γενικό νόμο με τον ειδικό νόμο, lex specialis και lex generalis. Νομίζω ότι lex specialis μπορεί να δικαιολογηθεί μονάχα σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κάτι τόσο ιδιαίτερο, κάτι τόσο συγκεκριμένο, τόσο εξειδικευμένο, το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί κανονιστικά με διαφορετικό τρόπο η γενική ιδέα ότι όλα αυτά τα σώματα, οι βρίσκονται ε, και οι αρχές ε, ε, θα βρίσκονται κάτω από μια γενική ομπρέλα βεβαίως είναι καλοδεχούμενο σαν αρχή. Υπάρχουν ε, και κάποιες ε, διασφαλίσεις ε, οι οποίες δεν ήταν παρούσες στις ρυθμίσεις για την δικαιοσύνη και την αστυνομία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε γενικούς κανονισμούς που ήδη να αναγνωρίζουν τις πιο υψηλές αρχές και για ορισμένες περιπτώσεις να προβλέπονται ακόμα πιο υψηλά πρότυπα, πιο υψηλά στάνταρ. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να γίνουν με τη σωστή χρονολογική σειρά γιατί ε, το timing είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάνω από 60 σώματα και θεσμικά όργανα και λοιπά που ε, θα πρέπει να ε, συνδυαστούν. Privacy Shield. σε μερικές ώρες, αυτή τη βδομάδα, εν πάση περιπτώσει, επίκειται πριν και φύγουμε για την ε, Washington DC, προβλέπεται η ανακοίνωση η οποία θα αναφέρεται ακριβώς στις πρόσφατες εξελίξεις στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, τροποποιήσεις ε, ε, της πράξης για τις θεωρήσεις, Visa Act κλπ και επίσης θα προσθεθούν και κάποιες νέες σκέψεις επί τη βάση των όσων συμφωνήσαμε με τους συναδέλφους των Εθνικών Αρχών με την ευκαιρία της, ε, σωστής, ε, της ε, πρόσφατης συνάντησής μας. τα παρατήματα ε, του Protection Shield είναι μοναδικά σε ολόκληρο τον κόσμο ε, και βεβαίως ε, η προσπάθεια συλλογής πληροφοριών intelligence θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σωστό και η χρήση των δεδομένων Privacy Shield είναι ένα από αυτά τα θέματα και εάν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει και να έχει τα ωφέλη της μεταφοράς των εμπορικών δεδομένων θα πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστεί ταυτόχρονα τις ε, βασικές ε, αρχές. Όσον αφορά τα θέματα αυτά εμείς τα προσεγγίζουμε με αρχές διαφάνειας, ωστόσο πιστεύουμε ότι δεν έχουμε φτάσει στο σωστό ε, επίπεδο και θα πρέπει οπωσδήποτε τα διδάγματα, να εξάγουμε διδάγματα από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καθορίζουμε επομένως ε, τις, ε, ε, τα πεδία τα οποία εξακολουθούν να είναι σημαντικά, κυρίως όσον αφορά την εποπτεία, την επιτήρηση. Έχουν, προβλέψει, έχουν προκύψει βεβαίως και κάποιες θετικές εξελίξεις όσον αφορά τα εμπορικά δεδομένα. Το Protection Shield δεν ήταν η κύρια προτεραιότητα για τις ΗΠΑ, ωστόσο ε, νομίζω ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε και βελτιώσεις μπορούμε να επιφέρουμε έτσι ώστε να αποφύγουμε, να ξαναδούμε ιστορίες που είδαμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουταρέλη, λέει η Πρόεδρος, για όλες τις παρατηρήσεις σας. Και βεβαίω σα ευχόμαστε καλή τύχη όσον αφορά τι νέε προκλήσει που έχετε μπροστά σα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σα εδώ, τη συζήτηση, τα πολύ ενδιαφέροντα που μα είπατε. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει 26 Μαρτίου και την επόμενη μέρα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.